Να ενημερώσω επίση το Κοινοβούλιο ότι σύμφωνα με τον κανόνα 231 παράγραφος 4 δεν εκφράστηκε έτοιμα να ψηφιστεί το διορθωτικό που αναγγέλθηκε χθε στις 5 το απόγευμα και λοιπόν το διορθωτικό εγκρίνεται. Τέλος.